Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους και τον υποψήφιο επίτροπο για τις απαντήσεις του. Και τώρα, κύριε υποψήφιο επίτροπε, έχετε χρόνο για μια καταληκτική απάντηση που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το πεντάλεπτο. Μπορείτε να πάρετε και δύο λεπτά παραπάνω αν χρειαστεί από το χρόνο μας, διότι υπήρξατε ιδιαίτερα πειθαρχημένος. Οπότε Εάν θέλετε, θα μπορούσατε να επανέλθετε και σε κάποιο ερώτημα ή απάντηση που δεν είχατε χρόνο να απαντήσετε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την καταληκτική σας ομιλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και σας Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την ε, τόσο καλή διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. Ελπίζω να είχατε την ε, αίσθηση ότι μπορέσατε να θέσετε τις ερωτήσεις που σας ενδιέφεραν. Ήταν ε, δίκαιη η ακρόαση όπως μου είχε περιγραφεί, αυτό και αισθάνθηκα, αλλά ελπίζω και εσείς να ρωτήσατε αυτά που θέλατε να ρωτήσετε. Σημειώνω ότι επαναλαμβάνονταν ε, στο περιεχόμενο τους κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια, θα τα μελετήσω με προσοχή και θα επικεντρωθώ σε κάποιους τομείς όπως και υποσχέθηκα. Ως προς το χαρτοφυλάκιό μου, θα ήθελα να ε, θυμίσω τις βασικές προτεραιότητες, αυτά που ελπίζω να πετύχω και που ελπίζω ότι συνδυάζονται με πολλά από αυτά που και εσείς αναφέρατε. Πρώτον, στον στο επίπεδο τη υλοποίηση θα πρέπει να συμπληρωθεί το έργο του προκατόχου μου και τη Επιτροπής σα, ώστε να υπάρξει σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Από την πρώτη μέρα θα αφοσιωθώ με ιδιαίτερη σπουδή στο να γίνει η Τραπεζική Ένωση, το CRD4 και το MIFID πραγματικότητα σε όλους τους τομείς. Έχω την εντύπωση, μια εντύπωση που αποκομίζω από τη συνάντηση αυτή, είναι ότι η πλειονότητα θέλει να ολοκληρώσω το έργο αυτό και θέλετε και το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ενεργά στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι ακριβώς και η δική μου πρόθεση. Υπάρχει ένα θέμα επιβολής αξιολόγησης και αποτίμησης και αναθεώρησης. Νομίζω σωστά το αναλύσαμε αυτό προηγουμένως. Δεν χρειάζονται κοινοί κανόνες εάν δεν τους ελέγχουμε και τους εφαρμόζουμε σωστά, αλλά πρέπει και να τους αναθεωρούμε εφόσον χρειάζεται. Νέες πηγές κινδύνου θα πρέπει και αυτές να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Μερικές ήδη αντιμετωπίζονται, όπως οι διαθετικές αλλαγές της τράπεζας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικά μεγάλες τράπεζες που κινδυνεύουν με πτώχευση, αλλά και άλλες, άλλοι τομείς όπως η εξωτραπεζική εξυγίανση. Κάτι που θα μας απασχολήσει και στο επίπεδο του G20. Στο διεθνέ επίπεδο τώρα. Ε, υπάρχει μια σαφής άποψη από την Επιτροπή σας ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι κανόνες εφαρμόζονται με τον ίδιο άψογο τρόπο και με ταχύτητα σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διεθνή συμπεφωνημένα πρότυπα για, με κοινού λογιστικούς κανόνες και ε, συγκεκριμένους δείκτες ε, συγκριτικής αξιολόγησης σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο κέντρο των διαπραγματεύσεων TTIP. Σε ό,τι αφορά καταναλωτές Υπήρξαν πολλές παρατηρήσεις για τη σημασία των καταναλωτών και των χρηστών των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπό την έννοια ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους καταναλωτές ως χρήστες, ως τελικούς δικαιούχους αυτών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συμφωνώ απολύτω. Θα πρέπει οι ενώσει των καταναλωτών να συμμετέχουν, να καταλάβουν γιατί προσπαθούμε να λειτουργήσει καλύτερα η κοινή αυτή η αγορά. Το ίδιο και για τι ασφαλιστικέ, το ίδιο και για την τράπεζα για, το, για τις τραπεζικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Ε, ελπίζω ότι θα πετύχω τη συνεργασία με την Επιτροπή σας και στον τομέα αυτό. Και κάτι ακόμη που τέθηκε είναι η σημασία των θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη απειλή κατά της σταθερότητας και νομίζω ότι η σταθερότητα ενδιαφέρει πολλού εδώ από ό,τι κατάλαβα. Η μεγαλύτερη απειλή κατά τη ε, σταθερότητα είναι η ψηλή ανεργία και η μηδενική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε κανονισμού ασχέτως με τους στόχους μας για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι υπό την αιγίδα της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών θα πρέπει να προπλέψουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για υπηρεσίες που κοινώς θα απευθύνονται και στα 28 κράτη-μέλη δημιουργώντας ε, δυνατότητες θέσεων εργασίας. Και το τονίζω αυτό και για τους 28. Θέλω να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε τις σχετικές προτάσεις μαζί. Και βραχυπρόθεσμα θα ε, δοθεί έμφαση, όπως μου ζητήθηκε και από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, να προωθηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα που ήδη έχει προβλεφθεί και το χρηματοπιστωτικό σύστημα να διδαματίσει το ρόλο του. Και τέλο, ένα άλλο μεγάλο θέμα που προέκυψε και από την άποψη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και σε κάτι που με αφορά προσωπικά. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με την διαφάνεια. Νομίζω ότι ω έννοια η διαφάνεια είναι κεντρική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αλλά είναι το ίδιο καθοριστική και για τη σωστή σχέση που ελπίζω να έχω μαζί σα. Ε, μπορεί από καιρού εις καιρό να διαφωνήσουμε σε κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ποτέ ε, στο ότι δεν πέτυχα αποτελέσματα που εσείς επιθυμούσατε ως προς τον αμοιβαίο σεβασμό και την διαφάνεια και τον ανοιχτό μας διάλογο. Ελπίζω ότι υπήρξα σαφής κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν πραγματιστή υπέρ της συνένεσης και ευρωπαϊστή, φιλευρωπαϊστή πολιτικό. Δεν είμαι ένας μεγάλος ρήτορας όσο είμαι κάποιος που αγαπά την δράση. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα όσα πέτυχα τα πολιτικά πράγματα, τα πέτυχα, διότι συνεργάστηκα με τους άλλους, είτε με τους συνεργάτες μου, δημόσιου υπαλλήλου, είτε με συναδέλφους και με ομολόγους μου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κομμάτων. Εφόσον με εγκρίνετε με το ίδιο πνεύμα θα συνεργαστώ και με όλους εσά. Νομίζω ότι εν είδη συμπεράσματος όλοι μας έχουμε πολύ σοβαρή ευθύνη να αναλάβουμε σε αυτή την κρίσιμη καμπή στην ιστορία της Επίρου μας. Νομίζω οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν αλλάξουν προς το καλύτερο. Και νομίζω ότι από κοινού στον τομέα αυτό μπορούμε να διδραματίσουμε έναν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία. αναμένω λοιπόν και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σα για να φέρω ει πέρα σε αυτά τα καθήκοντα, να μπορέσουμε από κοινού να έχουμε έναν κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που να είναι διαθετημένο σωστά, να λειτουργεί προς το συμφέρον όλων και να δίνει ε, το, ε, να επιτρέπει να κυλά το αίμα στις φλέβες ενός οικονομικού κλάδου που θα προσφέρει ωφέλη σε όλους, στους πολίτες. Και ότι θα ανακτήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εμά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε πραγματικά να ριζώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καρδιά τους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε υποψήφια επίτροπε και τώρα Έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών για να γίνει αξιολόγηση της, ακριο... της ακρόασης από τις 5.30 μέχρι τις, 5... 7. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Σάρον Μπόουλς, η οποία ήταν προκατοχός μου εδώ πέρα στην Προεδρία και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Γεια σου Σάρον, τον Τζόναθαν Χίλ να ευχαριστήσουμε και όλους σας πέρα στις συνεδρίες σας.